E, Καλή σας μέρα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την συνεδρίαση. Κυρίες και κύριοι, θα ήμουν ευγνώμων αν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε. Chciałbym że otrzymałem pismo od przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana. Και καλώς ήρθατε. Και έχουμε και επιστολή του κυρίου Φαν Ρόμποϊ που μας ενημερώνει για την απόφαση του Συμβουλίου σε σχέση με τις διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο